Τελευταίο σημείο τη ημέρα διάταξη, η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το αρχιπέλαγος των Σβάλμπαρντ και ε, του αλληλευτικού πόρου του αρχιπέλαγους. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Βαλέζα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν ήρθε η αρμόδια επίτροπο Αλίες ε, η κυρία Δαμανάκη, αλλά ευχαριστούμε εκ μέρου τη Επιτροπή Αλίε για τη δυνατότητα που μα δίνετε. Και χαίρομαι που δίνουμε την ευκαιρία για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νομικό Καθεστώ του αρχιπελάγου Σβάλμπαρτ και των αληφτικών αποθεμάτων του. Η ερώτησή μα αφορά ε, ένα επικίνδυνο πρόβλημα που ανέκυψε τα τελευταία χρόνια και τι τις ποσοστώσεις ε, του, της υπόγλωσσας της Γρυλανδίας στην περιοχή του ε, Σβάπαλτ. Γιατί το αρχιπέλαγο Σβάπαλτ έχει εκχωρηθεί στην Νορβηγία με τη συνθήκη της Πιτσφέργης που διασφαλίζει νομικό καθεστώς ισοτιμίας για την περιοχή Πράγμα που περιλαμβάνει και την αρχή της καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταπολέμηση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους αλληλευτικούς πόρους του αρχιπελάγου Σβάλμπαρτ. Το 1977 η Νορβηγία ανακήρυξε μόνο μερός το αρχιπέλαγος ζώνη προστασίας της αλίας του Σβάλμπαρτ και ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις της συνθήκης της Σπιτσμπέργκης κατά των διακρίσεων δεν ισχύουν σε αυτή τη ζώνη. Το 2010 η Νορβηγία και η Ρωσία υπέγραψαν στο Μούρμανσκ συνθήκη θαλάσσιας οριοθέτησης σχετικά με τη θάλασσα Μπάρεντς. Ορισμένα από τα ύδατα της ζώνης προστασίας αλίας του Σβάλμπαρτ βρίσκονται σήμερα ανατολικά από τη γραμμή οριοθέτησης, τη γραμμή Μούρμανσκ. Η Νορβηγία και η Ρωσία συνεργάζονται στα πλαίσια της μικτής Νόρβηγο-Ρωσικής Επιτροπής Αλίας για τη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων στη θάλασσα Μπάρινς. Τα τελευταία χρόνια αυτό οδήγησε στον σφετερισμό αλληλευτικών δυνατοτήτων, προζημίαν μάλιστα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα όσον αφορά την Ορβηγία. Γιατί η λήψη ενωσιακής δράσης, η Νορβηγία θα διαθετεί όλα τα ζητήματα ανάλογα με το συμφέρον της. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω μερικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρη της συνθήκης της Σπιτσβέργης του 1920 απολάβουν ίσων δικαιωμάτων ως προς την αλληλεία στη ζώνη προστασίας αλίας του Σβάλμπαρτ. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με το νομικό καθεστώς του τμήματος της Ζώνης Προστασίας αελίας ανατολικά της γράμμης Μούρμανσκ. Θεωρείτε ότι αυτό το τμήμα εμπίπτει στα διεθνή ύδατα πάνω από τη ρωσική υφαλοκρηπίδα ή είναι πλέον μέρος της ρωσικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τρίτη ερώτηση. Αν οι ελίς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χάσει το δικαίωμά τους να αλλιεύουν στη ζώνη προστασίας αλίας ανατολικά της γραμμής Μούρμανσκ στο αρχιπέλαγος Βάλμπαρτ. Εξετάζει η Επιτροπή το δεχόμενο να ζητήσει αποζημίωση. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με την νομιμότητα της μεταφοράς από την Νορβηγία στη Ρωσία της ευθύνη για μέρος της νορβηγικής ε, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στη θάλασσα του Μπάρεντς. Και πέμπτη και τελευταία ερώτηση. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέρος στη συνεδρίαση της μικτής Νορβηγο-Ρωσικής Επιτροπής Αλληλείας που θα γίνει το 2014 ή σε άλλες συνεδριάσεις ώστε να αποφευθεί η παράνομη ιδιοποίηση ποσοστώσεων επί της υπόγλωσσας της Γρυλανδίας και του κοκκινόψαρου ε, ή του πλάτακα στη θάλασσα του Μπάρεντς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος ο κ. Ποτότσνικ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να απαντήσω στο όνομα της συναδέρφου μου, της Επιτρόπου Δαμανάκη, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα στη σημερινή συνάντηση. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα, που επέστησε την προσοχή μας στα σημαντικά αυτά ερωτήματα. Επιτρέψτε μου να τονίσω πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό που συνδέεται με την αλληλεία. Αφορά πολύ λεπτές στοιχές του διεθνούς δικαίου. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι συνδέεται με τις σχέσεις μας με την Νορβηγία, που και τώρα αλλά και στο παρελθόν ήταν ο πιο σημαντικός εταίρος μας στην αλληλεία και σε άλλα θέματα που συνδέονται με τη θάλασσα, μεταξύ άλλων ε, θεμάτων της Ακτικής. Ήταν ε, πάντα θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έχουν συνυπογράψει την ε, συνθήκη του 1920, τη συνθήκη της ε, Σπιτσβέργης, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη της συνθήκης αυτής. Όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης της αλληλείας και την αποδοχή μέτρων που προτείνει η Νορβηγία σχετικά με τα ύδατα γύρω από το Σφάλβαρτ εφαρμόζονται με τρόπο μη διακριτικό ε, και βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές και επίσης γίνονται σεβαστά από, από όλους τους ενδιαφερομένους. Όσον αφορά τις σε 3 και 4 του ε, Ευρωβουλευτή, δεν υπάρχει θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά. Οι συνέπειες ε, της γραμμής του Μουρμάνσκ για την αλληλεία στα ύδατα αυτά εξετάζεται ακόμα σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει τις ε, διαδικασίες ε, της ε, κοινή Ρώσο-Νορβηγικής συμφωνίας. Είναι διμερή συμφωνία και δεν αποτελεί περιφερειακή ρύθμιση της αλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να συμμετέχει στις σχετικές συναντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει να έχουν πάρθει ποσοστό όσον αφορά την υπόγλωσσα τη Βλανδία και του κοκκινόψαρου στην περιοχή. Έτσι λοιπόν δεν έχει γνώμη για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στου αγορητέ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, ξεκινώντα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Φράγα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βαγουένσα για την πρωτοβουλία του προκειμένου να μην πέσουν στη λύθη τα αλληλευτικά μας δικαιώματα στο Σβάλπαρτ. Ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν έχει διευκρινιστεί, όπως είδαμε και σήμερα το βράδυ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Ελευτικής Συμφωνίας με την Ορβηγία, αν σε αυτές ο, δια, ο διαπραγματευτής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε συζήτηση ή διαπραγμάτευση προκειμένου να βελτιωθούν οι αλληλευτικέ συνθήκες τη παρεμπίπτωσης της Ελίας Εγκλεφίνου στο Σβάλπαρτ και να απαλλαγούμε από τις ε, παρεμβάσεις της Νορβηγίας στην αλήψη των ποσοστώσεων γάδου. Ε, ενώ σε αντάλλαγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραιτηθεί από άλλα αλληλευτικά της δικαιώματα. Είναι ένα μείζο ζήτημα γιατί όσο ευπρόσδεκτες και αν είναι οι βελτιώσεις, μένουν στον αέρα άλλα πολύ σημαντικά δικαιώματα άλλων αλληλευτικών στόλων. Και δεδομένου ότι μέχρι στιγμή ε, και οι ενδιαφερόμενε χώρε όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζουν την άποψη ότι η ερμηνεία που κάνει η Νορβηγία τη συνθήκη των Παρισίων και οι συνέπειε ε, τη δημιουργία ζώνη προστασία ελεία αντίκειτο στο διεθνέ δίκαιο και στο δίκαιο τη θάλασσα, θα ήθελα να μάθω από πού ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τη διαπραγμάτευση του των, ε, των μελλοντικών μα ποσοστώσεων στο Σβάλμπαρτ ποιοι ήταν οι όροι αυτής της προσφοράς και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συζητήσει το θέμα αυτό πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη και αν είχε συγκεκριμένη εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η διάλεκτη συμπεριφορά της Νορβηγίας στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει, δεν έχει υπογράψει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Θήκη των Παρισίων. Οπότε θεωρεί ότι μόνο με τα κράτη-μέλη η Νορβηγία θα έχει διαπραγματεύσει. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμποδίζει τα κράτη-μέλη να έχουν διμερεί διαπραγματεύσει με την Νορβηγία, θεωρώντα ότι αυτό το θέμα εμπίπτει στι αποκλειστικέ αρμοδιότητε. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι δύο αυτέ απαντήσει. Τι συνέβη στι πρόσφατε διαπραγματεύσει με την Νορβηγία, γιατί έμεινε εμβρόντιτο και ο ελευτικό κλάδο, αλλά και τα κράτη-μέλη από τι διαπραγματεύσει αυτέ. Σας ευχαριστώ για την Άλντε. Το λόγο έχει ο κύριος Γκάλαγκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν θέσει το ζήτημα και όσον αφορά το θέμα της Αρκτικής και θα πρέπει να δούμε να πούμε ότι έδωσε ειδική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Νορβηγία ούτως ώστε να έχει καθεστώς παρατηρητού στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Υπάρχει επιστημονική συνεργασία εντυπωσιακή όσον αφορά την περιοχή αυτή, κυρίως στον τομέα της έρευνας για την αλλαγή του κλίματος και το περιβάλλον και όλα αυτά στην περιοχή Σβάλμπαρτ. Και είχα τη δυνατότητα να το δω με τα ίδια μου τα μάτια όταν έκανα επίσκεψη εκεί πέρυσι τον Ιούνιο. Και θα πρέπει, είδα δυνατότητα να δούμε την απώλεια πάγου στην περιοχή και έγιναν πιο προσβάσιμες οι λευτικές περιοχές τότε. Λοιπόν, και το θέμα λοιπόν των αλληλευτικών δικαιωμάτων στον τομέα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε και ποια είναι η νομική κατάσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν και διευκρινίσεις από την νορβηγική κυβέρνηση, ούτω ώστε να μην υπάρχει διακριτική αντιμετώπιση των κρατώμελων μελών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο αρχιπέλαγο Σβάλμπαρτ. Τώρα φαίνεται ότι είναι καλή στιγμή να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η νορβηγική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Σάλμπεργκ ε, θέλει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει συνεργασία Νορβηγίας-Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ανέφερε η κυβέρνηση ότι προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τι σχέσει και του δεσμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νορβηγία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη επιτυχώ συνεργάζονται και έχουν κοινή διαχείριση ελευτικών πόρων στο Βόρειο Ατλαντικό και θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου τον συνάδελφο Βαλέσα που μα έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που απάντησε εκ μέρους της Επιτρόπου της Υπευθύνου για τα θέματα Λίας. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Η κυρία Λοβίν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τον Σεπτέμβριο του 2012... Ο πάγος στην Αρκτική ε, είχε τη μικρότερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ από δορυφόρους. Ήταν περίπου το μισό από ότι το ελάχιστο από το 1981 μέχρι το 2010. Ο πάγος ε, καλύπτει σημαντικό μέρος ε, της ε, θαλάσσιας ζώνης γύρω από το Σφάλμπαρτ το συνήθως, αλλά τώρα αυτό αλλάζει. Μπορείτε να δείτε πόσο λιώνουν οι πάγοι με τρομακτική ταχύτητα και ανοίγουν νέοι δρόμοι για μεταφορές, εξόριξη πετρελαίου, αερίου και αλία ανάλογα με τις διάφορες ερμηνείες ε, της ε, συνθήκης ε, του 1920 δεν με εκπλήσει η πρωτοβουλία να έχουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των αλλιευτικών κρατών αλλά η περιοχή εκεί. Ε, επί 800.000 χρόνια δεν ήταν προσβάσιμα τα νερά κάτω από του πάγους και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη προτού να είναι πολύ αργά να προστατεύσουμε αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Η Νορβηγία, όπω ε, συμβαίνει συχνά, ε, παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη βδομάδα, πραγματοποιείται μια συνάντηση στη Γρυλανδία ανάμεσα στα πέντε κράτη της Ακτική. Ο Καναδά, η Δανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να πείσουν τη Ρωσία και την Νορβηγία να ε, έχουν απαγόρευση αλίας ε, στην Αρκτική, κάτι, ε, το οποίο δεν έχει, κάτι για το οποίο δεν έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα η Νορβηγία, κάτι που δεν με εκπλήσει. Η Νορβηγία είναι χώρα γειτονική με τη δική μου χώρα, την Σουηδία, αλλά οποιαδήποτε οποιοδήποτε ισχυρισμός της Νορβηγίας για να ληφθεί σοβαρά θα πρέπει να σημαίνει ότι η Νορβηγία θα πάρει το πλευρό όχι της Ρωσίας αλλά των άλλων κρατών. Δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ε, την περιοχή αυτή, καλύτερα να την αφήσουμε όσο έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πατράου Νέβες έχει λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε το νομικό καθεστώς και πρόσβαση στου αλληλευτικούς πόρους του αρχιπελάγου Σβάλμπαρτ, όπου μονομερός η Νορβηγία ανακήρυξε ζώνη προστασίας αλληλεία, που εν μέρη περιλαμβάνεται στο, στη συνθήκη οριοθέτησης της θάλασσας του Μπάρες που συνήψε με την Ρωσία απαιτεί άμεση αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ένομα συμφέροντα των αλληλευτικών στόλων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Για μία ακόμη φορά, η χρήση των δικαιωμάτων αλλία, η εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων και ο σφετερισμό αλληλευτικών πόρων και κοινών αλληλευτικών πόρων έγινε προς όφελος τρίτων χωρών και εις βάρος των συμφερόντων των ε, χωρών μελών. Όπως διαπιστώσαμε και σε άλλες περιπτώσεις, τέτοια μέτρα που λαμβάνονται από τρίτες χώρες εις βάρος ε, ε, των πολυμερών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σημαντική απειλή της ισορροπίας των ελευτικών πόρων, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ελευτικού κλάδου, δημιουργώντας στρεβλώσεις εμπορικές και αθέμητο ανταγωνισμό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων. Ε, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και πολύ σοβαρή και απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και ανάλογα μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή να είναι περιοριστική, προστατευτική και υπερβολική, υπερβολικά απαιτητική σε εσωτερικό επίπεδο, να είναι χαλαρή, επίκη ε, και διαλλακτική σε εξωτερικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και μάλιστα κατάλληλα και αποτελεσματικά για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους και η βιωσιμότητα του ελευτικού κλάδου. Ως πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει στην επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Αλληλευτικής Επιτροπής Ρωσίας-Νορβηγίας ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να, να προασπίσει με πυγμή και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ένομα συμφέροντα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Στόλου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητηθεί να μιλήσει κανείς στη δικασία Catch Δίνω λοιπόν το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Ποτότσνικ. Thank Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτές, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι γνωρίζουμε τη συνθήκη του Μουρμάνσκ που ε, έχει συνάψει η Νορβηγία με την Ρωσία το 2010 και που έχει οδηγήσει και που έχει κλείσει τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρε αυτέ ε, όσον αφορά την οριοθέτηση ε, τη θάλασσα Μπάρεν. Αυτό βέβαια μπορεί μόνο να ωφελήσει την πολιτική στην πιο ευαίσθητη αυτή ακτική περιοχή. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει αν η γραμμή οριοθέτησης έχει αρνητικέ συνέπειε για τα σκάφη τη Ένωση που αλλιεύουν στην περιοχή και ε, αν είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα στην ε, Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τον νόμο της θάλασσας. Επίσης, ε, θέλω να επαναλάβω ότι όσον αφορά τις ποσοστώσεις, δεν γνωρίζουμε να ε, υπάρχει κάποια απαλωτρίωση των ποσοστώσεων υπόγλωσσας της Βιλανδίας και του κοκκινόψαρου στην περιοχή. Η κυρία Φράγα Στέβες έθεσε μια ερώτηση και μπορώ να πω μόνο ότι είναι πολύ αναλυτικές αυτές οι ερωτήσεις. Δυσκολεύομαι να απαντήσω, αλλά σίγουρα θα τις μεταφέρω στην συνάδελφό μου και θα φροντίσω να απαντηθούν. Τέλος, θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας. Στην δήλωση τις ε, συναδέρφους σας ε, από τους Πρασίνους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της βιωσιμότητας της Αρκτικής και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος ε, είτε από άλλες πλευρές. Είχα επισκεφτεί το Σφάλμπαρτ πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να γνωρίζετε ότι υπάρχει εκεί περιοχή όπου συμμετέχουν πολλοί διεθνείς επιστήμονες. Είναι πολύ όμορφη περιοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περατώθηκε η συζήτηση. Η επόμενη σύνοδος θα λάβει χώρα αύριο 5η 27 Φεβρουαρίου 2014 από τις 8.30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη δημοσιεύτηκε και είναι διαθέσιμη στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε διακόπτεται η